Dear President, Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω τη συνεδρίαση. Έχουν διανεμηθεί τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν χτες. Παρατηρήσει έχετε. nicht der fall. Όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ακολουθεί η συζήτηση για έξι ψηφίσματα για τη Γουινέα και θα